Κένια. Λοιπόν, γνωρίζετε τη φράση που θέλω να πω για τα ψηφίσματα αυτά και τώρα θέτω σε ψήφιση ε, με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Ψήφισαν 47, 46 υπέρ, κανείς κατά, μία αποχή εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία. Έκλεισε με τις ψηφοφορίες, η, τα πρακτικά θα υποβληθούν στην ε,